και επί των οποίων, εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, θα επιφέρουμε πάρα πολλέ βελτιώσει στην ισχύουσα νομοθεσία. Ε, υπάρχει μια κέντρο κατευθυνόμενη διαδικασία η οποία ε, έχει να κάνει με αυτή τη διαδικασία της έγκρισης και ταυτόχρονα να υπάρχει ασφάλεια διατροφής πριν τη θέση εμπορία, ετικετοθεσία για όλα τα συστατικά και τις πρώτες ύλες. Απλουστευμένη διαδικασία σε σχέση με τα παραδοσιακά από τρίτες χώρες και η διευκόλυνση προσβασιμότητας αγορές. Επίσης, ε, θα πρέπει και οι εμπορευόμενοι να ε, κοινοποιούν το ότι υπάρχει, έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα από ζώα που έχουν υποστεί πειράματα. Επομένως, θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς να κάνουμε κανένα συμβασμό όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια να μπορέσουμε να συνοηθούμε και αμελητή να προβούμε στις απαραίτητες βελτιώσεις νομοθεσίας ούτως ώστε να υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες ε, ε, βελτιώσεις όσον αφορά την κοινοτομία αλλά και τον κλάδο της, ε, των διατροφής. Επομένως, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε επομένως, να δώσουμε μια όθηση στις διαπραγματεύσεις και θα βρεθεί κάποια διέξοδο σύντομα. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, εάν δεν μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα, αυτό συνέβη παρά ότι έχουμε κάποια θετικά βήματα όσον αφορά την κλωνοποίηση κατά αυτές τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και εμείς ε, διατηρούμε τη δέσμευσή μας ώστε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις ε, κατόπιν του Οκτωβρίου 2010. Και σας προτείνω τα εξή. Προσωρινή αναστολή της χρήσης κλωνοποίησης και αναστολή των εισαγωγών τέτοιων προϊόντων και να υπάρχει σύστημα ανιχνευστημότητας όσον αφορά έμβρια και σπέρμα από κλωνοποιημένα ζώα. Αναγνωρίζουμε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο κατά τη διαδικασία τη συνδιαλλαγή. Επίση, σαφώ προκύπτει το ότι για την κλωνοποίηση θα πρέπει να βρεθεί κάποια συμφωνία και να ισχύσει αναλογικότητα και να σας υποβάλουμε μετά την αξιολόγηση μια ολοκληρωμένη πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχει συμφιλιωτική νοοτροπία ο κύριο Επιτέλου αλλά και η Προεδρία. Θα πρέπει να κάνουμε τα επόμενα βήματα και εγώ προτίθεμαι να συνεχθώ μαζί σα αλλά και με το Συμβούλιο όσον αφορά ενδεχόμενα σενάρια ε, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα και να συμφωνήσουμε πάνω σε μια διαδικασία που θα μα οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να γίνει προβληματισμό από όλε τι πλευρέ για να μπορέσουμε να πάμε καλά ε, και στα δύο υποζήτηση ζητήματα, ούτω ώστε όλο ο κόσμο να ωφεληθεί και τώρα. Οι αγορητέ των πολιτικών ομάδων. Για δύο λεπτάκια για το Λαϊκό Κόμμα, κυρία Αγιούσο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, το πρώτο θέλω να πω είναι να συγχαρώ την κυρία Λιωτάρ, την Προεδρία και τον Επίτροπο και το Επιτελείο τους διότι κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες δυστυχώς όμως πρόκειται για ένα σημαντικό κανονισμό που χρειάζεται αλλά δεν είχε ο τέλος αυτή η υπόθεση ε, σε σχέση με αυτά τα οποία θέλουμε ε, να, να, να, να ορίσουμε για την αιτιοδοθεσία που δεν είναι ρεαλιστικά. Ε, χρειάζεται ρεαλισμός όσον αφορά το τι θα προβλέπει για τα συστατικά. Χάθηκε μια ευκαιρία να μπορούσαμε να κάνουμε πώ θα εμπρό ο σχετικός ε, κλάδος για, τα, για, τα, είδη διατροφής τώρα έχει ως φραγμό στην προδό του αυτήν την ε, αρχαϊκή και απαρχιωμένη νομοθεσία. Επιβάλλουμε γραφειοκρατία, ε, βαραίνουμε πάρα πολύ τον κλάδο. Δεν θα πρέπει επομένω να αυτά να τα επιβάλλουμε και σε τρίτους. Δεν είναι δυνατόν επίση να θεσπίζουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε γιατί έτσι εξαπατούμε του καταναλωτέ να συμφωνήσουμε. Πρόκειται για έναν κανονισμό που δεν αφορά μόνο, τον, μόνο την, την κλωνοποίηση, αλλά αφορά και άλλα ζητήματα. Η διατροφή από τρίτες χώρες και είναι και άλλα θέματα τα οποία και τα συμφωνήσαμε και έχουν σημασία τους καταναλωτές και για την εσωτερική αγορά αλλά και από πλευράς καινοτομίας και πολιτικής υγείας. Επομένως, ας πάρει αυτά τα θέματα τα πιο επίμαχα και ας τα κάνει χωρίς την πρόταση η Κομισιόν και να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε ό,τι θέλουμε όσον αφορά ε, την κλωνοποίηση. Να λάβουμε υπόψη όλη την επιστημονική τεκμηρίωση. Η η Κομισιόν έχει δεσμευτεί εδώ, ενώπιόν μας. Ε, και γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι το του δυνατόν κάτι θα κάνει η Κομισιόν προ αυτήν την κατεύθυνση. Η Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Γιώργο και τώρα για του σοσιαλιστέ. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Λάινεν. Κυρία Πρόεδρε, κυρία ε, Πρόεδρε της, ε, του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχω συμμετάσχει σε πολλές διαδικασίες συνδιαλλαγής, αλλά από τι 7 το απόγευμα μέχρι 7 το πρωί προσπάθειες σε διαδικασίες συνδιαλλαγής νομίζω είναι άνευ προηγουμένου και θα μένουν για καιρό χαραγμένες στις, μήλες, μνήμες. Δείχνει πόσο μεγάλη σημασία ε, το σύνολο των εμπλεκομένων σε αυτήν την προσπάθεια στη σημασία στην ε, προστασία των δικαιωμάτων των ε, πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον αυτό προσπάθησε να προαγάγει την υγεία, την προσοχή των δικαιωμάτων των πολιτών, ενώ από την άλλη πλευρά βρέθηκε αντιμέτωπο με τα ους ε, εκπροσώπους και τα συμφέροντα τη βιομηχανία της ε, παραγωγή κρέατος. Νομίζω ότι μπορούμε να συγχαρούμε τον κύριο Πιτέλα και την ομάδα του, παρότι δεν κατέληξα σε αποτέλεσμα αυτή τη διαλλαγή. Και από εκεί και πέρα έρχεται η στιγμή να καλύψουμε το κενό. Κύριε Ντάλι, δύο είναι οι προτάσεις. Μία είναι αυτή που αφορά τα novel foods ε, και έχουμε συμφωνήσει ουσιαστικά για ένα κεντρικό σύστημα ε, πιστοποίηση για τι εισαγωγέ από τρίτα κράτη, για τα νανοηλικά και το δεύτερο ζήτημα που είναι η κλωνοποίηση. Έχετε ακούσει τι έχουμε πει όλοι μα ότι δεν θέλουμε τέτοια προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά ή μη τι άλλο θέλουμε σήμανση για να μπορεί να έχει την ελευθερία τη επιλογή ο καταναλωτή. Και πιστεύω ότι για την έτοιμο το Κοινοβούλιο θα καταθέσετε την πρόταση σας στο ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ κύριε Λάιρεν, η φιλελεύθερη τώρα η κυρία Λουπέζ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λεωτάρ και τον κύριο Πιτέλα και τον κύριο Λάινεν, όλη την ομάδα τη διαπραγματευτική που χάρη σε αυτήν έχουμε μια πολύ νέα θέση κατά τη διάρκεια αυτού του πολύ ε, μακρού διαλόγου και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Κοινοβούλιο ήταν ενωμένο για να υπερασπιστεί τη δημόσια υγεία και την υγεία του καταναλωτή και γι' αυτό έχουμε εκλεγεί. Δεν χρειάζεται να, τώρα βέβαια να ρίχνουμε ευθύνε από εδώ και από εκεί, αλλά να προχωρήσουμε μπροστά. Ωστόσο, τα γεγονότα μιλούν από μόνα του. Ε, όταν φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου το Κοινοβούλιο έχει ήδη υποχωρήσει σε πολλά θέματα,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 μπλοκαρίστηκε το θέμα. Αναρωτιόμασταν αν πρέπει να, ετικετο, να γίνεται ετικετοθεσία για τα προϊόντα που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά, αν και αυτό είναι κάτι το θεμελιώδες για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό που έγινε ήταν, ε, ε, είναι, απαράδεκτο, και είναι ε, μόνο προφάσεις όλα αυτά. Δεν επρόκειται ούτε για εμπορικό πόλεμο, ούτε για παραβίαση του ΠΟΕ. Από νομικής άποψης αυτό ήταν λάθος, ήταν ψέμα και από τεχνικής άποψης ήταν λάθος λάθο. Δεν θελήσαν να το κάνουν γιατί όπω είπε ο Γιώλαν πριν από λίγο ε, ε, δόθη προτεραιότητα σε άλλα συμφέροντα και όχι σε αυτά του καταναλωτή. Τώρα όμω πρέπει να προχωρήσουμε και γρήγορα. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί αυτή η υπόθεση τη κλωνοποίηση είναι ένα ακόμα στοιχείο που χρησιμοποιούν όλοι όσοι θέλουν να αμφισβητήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι ένα επιχείρημα μορφή απέναντι στα δικά μα όργανα. Είναι ένα επιχείρημα μορφή απέναντι στα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Καλό για όνομα του Θεού για αυτό το θέμα της κλωνοποίησης πρέπει να πάρουμε σαφή θέση γρήγορα για να απαγορεύσουμε όπως επιθυμούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και οι Ευρωπαίοι πολίτες την εμπορευματοποίηση κλωνοποιημένου κρέατος και των κατιόντων των κλωνοποιημένων ζώων. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Στίβενσον για ένα λεπτό. Πρόεδρε, μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειά, ο κανονισμός περί νέων τροφίμων κατέρευσε, στα εξών συνετέθη, γιατί δεν μπορούσε να βρεθεί συμβαστική λύση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, εγώ ή, ε, πραγματικά Είχα προειδοποιήσει για το ότι η πεισματική άρνηση ε, συμβιβασμού θα οδηγούσε σε καταστροφή. Τώρα χάσαμε σημαντική νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα. Η διαδικασία συνδιαλλαγής είναι σίγουρα ένας χρήσιμο μηχανισμός στην νομοθετική διαδικασία, αλλά είναι ε, άσκοπο και μάταιο αν οι συμμετέχοντε δεν είναι έτοιμοι να συνδιαλλαγούν και να συμβιβαστούν. Ε, εμείς ε, χρειαζόμαστε ε, ενημέρωση λοιπόν των κανόνων. Τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την οδηγία του 97 περί νέων τροφίμων που είναι τελείως ξεπερασμένη. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει στεναρό νομοθετικό όργανο το οποίο είναι περήφανο για τα όσα είχε επιτύχει μέσα μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας, πέρασε αυτό το στρες αντοχής. Τώρα η Κομισιόν πρέπει να υποβάλει νέα νομοθετική και ελπίζω πως οι ευρωβουλευτές θα μάθουν από τα σφάλματά τους και θα συνειδητοποιήσουν πως οι λαοί της Ευρώπης υποφέρουν αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπαρτιστάς για ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Λάινεν νομίζω εξέφρασε πολύ εύγλωτα την ε, κατάσταση. Βρισκόμαστε εδώ αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ των συμφερόντων της ε, βιομηχανίας του αφενό και της δημόσιας υγεία των δικαιωμάτων του καταναλωτή αφετέρου. Και νομίζω ότι εμεί μπορέσαμε να επιδείξουμε μια πολύ υπεύθυνη και σωστή στάση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορέσαμε ακόμη να δεχθούμε και ε, υποχωρήσει σε σχέση με τι αρχέ μα, αλλά δυστυχώ διαπιστώθηκε απόλυτη δισκαμψία από πλευρά του Συμβουλίου. Η ε, προσπάθειά μα για συμβιβασμό προσέχουν σε κλειστέ ε, πόρτε. Και μάλιστα ο επίτροπο Δεγκούχτα προσπάθησε κάποια στιγμή να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν τη αγνία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της Διαλλαγή ψευδεπίγραφα επιχειρήματα τάχα του, οργανισμού, ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου και αντίστοιχα τέτοια για να μας πείσει να υποχωρήσουμε. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, καταθέσει νέα πρόταση για τα novel foods. Υπήρχε μια σχεδόν ε, εξασφαλισμένη συμφωνία, αλλά χρειάζεται τώρα πλέον απόφαση για τα κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. Και κύριε Επίτροπε σας προειδοποιώ ότι πρέπει αυτό να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί ε, παόριστον ε, αυτό το ζήτημα. Πρέπει στην τωρινή μας θετία και όχι σε κάποια μελλοντική να ε, επανέλθει το θέμα. Εμείς πρέπει να επιληφθούμε στη διάρκεια της τρέχουσας θετίας για να καταλήξει αυτή η διαδικασία. Και τώρα η κυρία Λιωτάρ εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα θερμά να ευχαριστώ τους συναδέλφους μου ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Αντιπροσωπεία ε, στις διαδικασίες συνδιαλλαγές για την ομόφωνη υποστήριξη της οποίας έτυχα μέχρι τις τελευταίες ε, στιγμές των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την, το θαυμασμό μου για την πρέσβυρα της Ουγγαρίας η οποία έκανε ό,τι μπορούσε για να συμπράξει σε μια συμφωνία. Το ίδιο και ο κύριος Νταλή δεν τα καταφέραμε εν τέλει να συμφωνήσουμε. Όμως ο καταναλωτής είναι δυνατόν να αγοράζει προϊόντα ε, εν αγνία του ε, προϊόντα προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ενώ κατά 77% ε, οι καταναλωτές Ευρώπη τάσσονται κατά ε, τη διάθεση αυτών των προϊόντων στην αγορά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε να γίνει αυτός ο πόλεμος εις βάρος των καταναλωτών. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Μας είπαν κάποιοι από το Συμβούλιο, κάποιοι από την Επιτροπή ότι οι κανόνες του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου ε, μας υποχρεώνουν να δεχθούμε προϊόντα των κατιόντων αυτών των κλωνοποιημένων ζώων. Ο κύριος Δεγκούχτ ήρθε να μας ισχυριστεί κάτι τέτοιο, ενώ με κατάπληξή μου είδα σε ένα απόρριτο έγγραφο προερχόμενο από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου των Υπουργών ότι η απαγόρευση της κλωνοποίησης των κατιόντων ή μάλλον της διάθεσης κατιόντων κλωνοποιημένων ζώων ε, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν, δεν αντίκειται δηλαδή στους κανόνες ε, του ΔΟΕ και λέει ότι μια τέτοια απαγόρευση μπορεί να είναι σύμφωνη, σύνομη με τους κανόνες της, ε, του ΠΟΕ εφόσον ε, στόχο έχει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία τα συμφέροντα καταναλωτών. Ερωτώ λοιπόν, είναι ενήμερα για το έγγραφο αυτό της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου τα κράτη-μέλη. Και αν ναι, γιατί ακόμη μας μιλάτε για εμπορικό πόλεμο. Γιατί επισύεται αυτό το ε, σκιάχτρο ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία, ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι τη αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Εάν οι διαπραγματευτέ των κρατών μελών δεν είχαν δει το έγγραφο τη νομική σα υπηρεσία, θα ήταν σκάνδαλο βέβαια. Εάν το έχουν δει, γιατί να προβάλλονται ψευδεπίγραφα επιχειρήματα. Κύριε Νταλή, εσεί ω Επίτροπο, ω διαπραγματευτή εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είσαστε υποχρεωμένο να καταθέσετε νέε προτάσει. Στηριζόμαστε στη δική σα υποστήριξη και έρχομαι τώρα να δώσω το κείμενο στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Σα άφησα να ξεπεράσετε το χρόνο σα, μια ήταν εισηγήτρια. Η κυρία Λεπά, ένα να το λόγο. Πρόεδρε, είναι αδιανόητο αυτό που ακούσαμε από την κυρία Λιωτάχ. Επανέρχομαι λοιπόν με την ίδια ερώτηση, γιατί έχω μείνει κατάπληξη. Ερωτώ την Επιτροπή. Είχε και η Επιτροπή γνώση αυτή τη αυτής της πραγματογνωμοσύνης, αυτού του εγγράφου της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Είναι αδιανόητο επί εβδομάδες ολόκληρες να μα λέτε ότι κινδυνεύουμε με πόλεμο ανοιχτό σε επίπεδο ΠΟΕ. Ο κύριος Ντεγκιούχ να μα λέει ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε ούτε τα αεροπλάνα μα ούτε τίποτα εάν λάβουμε τέτοια απόφαση για απαγόρευση των κλωνοποιημένων και ενώ υπάρχει ε, πραγματογνωμοσύνη τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου που λέει Ακριβώ το αντίθετο. Θέλω απαντήσεις. Ε, η Πρόεδρος ε, βέβαια προ την ε, η συγγήτρια μόνο μπορείτε να απευθύνετε δυνάμει του κανονισμού ε, ερώτηση, αλλά βέβαια και ο Επίτροπος αν θέλει μπορεί να σας απαντήσει. Ο κύριος Ρώση έχει το λόγο παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω πως το Συμβούλιο ξεπέρασε τον εαυτό του. Αυτοί που εκπροσωπούν τους πολίτες είναι αυτοί που δημοκρατικά έχουν εκλεγεί από τους ίδιους τους πολίτες. Αν λοιπόν το Κοινοβούλιο συνέχισε να επιμένει στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια λέγοντα πως το κλωνοποιημένο κρέας δεν μας κάνει για τον κόσμο μας, για τους πολίτες μας, θα έπρεπε να το δεχτεί. Η ευθύνη για αυτή την επιλογή που είναι πολύ αρνητική για τη βιομηχανία είναι η ευθύνη το Συμβούλιο. Το κείμενο για το, για το κρέας του κλωνοποιημένου θα είχε εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Το Συμβούλιο δεν το θέλησε. Αυτό το ίδιο στο Συμβούλιο που από τη μια πλευρά λέει ότι πρέπει να απελευθερωθούν όλα ενώ από την άλλη μας επιβάλλει να αφαιρέσουμε το made in στα ε, προϊόντα υφαντουργίας γιατί δεν θέλει να δώσει τις σωστές πληροφορίες ε, για τον ε, καταναλωτή. Μας σπάει τα νεύρα αγαπητοί συνάδελφοι γιατί δεν θέλει να βάλει ετικέτες για να ξέρει ο κόσμος ε, τι τρώει. Όμω το Συμβούλιο και ευχαριστώ τον συνάδελφο Πιτέλα που κράτησε ψηλά την τιμή και τη βούληση όλων των Ευρωβουλευτών να απορρίψουν αυτήν την εκβιαστική πρόταση που ήθελε το Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω τον Πιτέλα, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους συναδέλφους που είχαν ε, το θάρρος ε, να μην κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω σε κάτι που στο οποίο πραγματικά πιστεύουμε πως ήταν χρήσιμο για τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ για τις ευχαριστίες, λέει η Πρόεδρος, και τώρα δίνω το λόγο στους άλλους ομιλητές, ο κύριος Λίζε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πίτρο Πενταλή, αγαπητοί συνάδελφοι. το λέω απογοήτευση, όντως. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι ευθύνεται για την αποτυχία η αντιπροσωπευτική η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι δεν θεωρώ πως είναι υπεύθυνη ούτε ο Επίτροπος ούτε η εδώ παρούσα Προεδρεύουσα. Άλλα ήταν τα όργανα, οι, οι φορείς του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνέβαλαν σε αυτή την αποτυχία ή πάντως στην ανυπαρξία συζητήσεως. Ο Επίτροπος De Kucht, επί παραδείγματι, αλλά και εκπρόσωποι των Υπουργείων ε, Οικονομικών από τη Γερμανία, τουλάχιστον ξέρω ότι επέσιαν ε, το σκιάχτρο ε, πολέμων εμπορικών, αντίστοιχων ε, με του πολέμου της Πανάνας και τέτοια φρικτά πράγματα, χωρίς όμως να είναι βάσιμα αυτά τα επιχειρήματα. Εχθές συζήτησα στο... Εχθές ε, ήρθε από το Βερολίνο ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στο Στρασβούργο ειδικά για να μου μιλήσει για το θέμα αυτό της πολιτικής για τα τρόφιμα. Τα επιχειρήματα λοιπόν του Αμερικανού εκπροσώπου δεν ήταν τόσο πιστικά ώστε να διαπιστώσω θα ήταν αδύνατο να βρεθεί συμφωνία. Του είπα ποια είναι η κατάσταση στην υπόθεση αυτή. Δεν φάνηκε λοιπόν να μην υπάρχει δυνατότητα για εξέβρεση συμφωνίας με τους Αμερικανούς. Εάν θέλαμε να βρούμε συμφωνία βέβαια. Εκεί όμως που εξεπλάγει πραγματικά είναι όταν οι Αμερικανοί, η Αμερικανική του μου έδωσε αυτό το έγγραφο που σας δείχνω ε, που είναι μια κατανομή των ε, οδηγιών για σήμανση προελεύσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κανόνες που ισχύουν δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε για το κιμά φεριπίν, για ένα πακέτο κοιμά χάμπουργκερ ή βιφτεκιού χάμπουργκερ πρέπει να καταγράφεται πάνω στο πακέτο από πού προέρχεται αυτός ο κιμάς. Τι μας λέτε λοιπόν ότι θα έχουμε πόλεμο εμπορικό εάν ζητήσουμε την σήμανση του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένο ή από κατιόντες ε, ή ε, από γόνους κλωνοποιημένων ζώων. Εφόσον και οι ίδιοι Αμερικανοί έχουν το σύστημα αυτό της σήμανσης της προέλευσης ζώου, γιατί δεν θα δεχθούν να εφαρμοστεί αυτό σε κάποιο άλλο κράτος. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Μακάβαν για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Είπατε για το αν κατηγορούμε κάποιον, αλλά ήρθε η ώρα επιτέλου να είμαστε κάπω ε, ειλικρινεί. Ε, συμφωνήσαμε για το, την κλωνοποίηση, αλλά είπαμε ότι να μην ε, τρώμε τα κλωνοποιημένα ζώα και υπήρχε αυτό το θέμα στι διαπραγματεύσει. Δεν μπορέσατε να κάνετε τίποτα όσον αφορά την εισαγωγή τέτοιων ζώων και όσον αφορά το, το σπέρμα των ζώων και επίσης τον ε, απογόνων ε, και επομένω έχουν πρωτοπλασιασμό που ξεκινάει από αυτά τα ένα ζώα. Πώ θα να υπάρχει νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την θέση σε εμπορία ε, παραπροϊόντων από γούνα, γάτα, φώκια και γενικά να αξιοποιούνται ζώα και παραπροϊόντα τους που προέρχονται από πειράματα. Άρα, να αντιμετωπιστεί ε, η κατάσταση αυτή όσον αφορά την κλωνοποίηση. Δεν είναι θέμα ΠΟΕ. Είναι θέμα πολιτική βούληση. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτό θα ικανοποιήσει και εμά ω Κοινοβούλιο και αυτό θα πρέπει να είναι το θεμέλιο επί το οποίο να προχωρήσει η συμφωνία. Κύριε Μακαβάνη, συμφωνούμε λίγο πρόεδρο και δίνω το λόγο στην κυρία Ρόσμπαχ για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Τεράστιο έργο επετέλεσε, κυρία Λιωτάρ, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, σημειώθηκε διαφωνία όσον αφορά τα είδη διατροφής που προέρχονται από ζώα χρονοποιημένα. Στη δική μου χώρα απαγορεύεται η χρονοποίηση. Όμως προϊόντα τέτοια μπαίνουν κατά κάποιο τρόπο από την Κερκόπορτα, μπαίνουν στη χώρα μας τελικά. Και επομένως θέλουμε να πρετανεύσει η διαφάνεια. Γιατί ενώ έχουμε για τηλεοράσεις, για, για, για, για χάπια, για ζάχαρη, ένας σωρό διατάξεις. Εδώ τι κάνουμε. Θα πρέπει να υπάρχει πάνω στην ετικέτα, στο πακέτο, στη συσκευασία, ενημέρωση του καταναλωτή. Ας κάνουμε περισσότερα για την υγεία μας, για τα τρόφιμα, για την κτηνοτροφία, γιατί θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες μας και έναντι ημών, αλλά και έναντι των παιδιών μας. Χασί, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς έχουμε διαφωνία, έχουμε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για αυτή την νομοθεσία. Καλά το είπαν οι συνάδελφοι ότι Επιτροπή και Συμβούλιο δεν θέλουν να δώσουν την προτεραιότητα τα σημεία τα οποία προκάλεσαν την προστριβή. Έτσι θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών για χάρη κάποιων οικονομικών συμφορώντων. Δεν γίνεται να έχουμε κρέας και γάλα, αποκλωμμένα ζώα και έτσι ε, έπρεπε κάτι να κάνουμε για αυτά τα ζώα τα οποία υποφέρουν θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Εσείς, εσείς να είστε γιατί το κοινοβούλιο έκανε πάρα πολλές παραχωρήσεις έκανε πίσω σε πολλές διατάξεις και όσον αφορά την συσκευασία. Λιωτάρ και η Λύσε οι συνάδελφοι αυτοί μας εξήγησαν τι ισχύει και καταλάβαμε ότι τελικά ήταν αναλυθείς αν οι θέσεις του Συμβουλίου. Εάν θέλουμε να κλείσει αυτή η υπόθεση αισίως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την επιθυμία του κόσμου. Δεν θέλουν τέτοιο, τέτοια, τέτοιο ε, ε, κρέας από τέτοια ζώα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια πρώτη γενική παρατήρηση. Όταν μιλούμε για ε, δυσπιστία του καταναλωτή εις βάρος ε, των ε, ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή καλύτερα για παραγνώριση της ε, δουλειάς τους ε, πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάμε ποιοι είναι αυτοί που παραγνωρίζουν τη δουλειά και τι αρμοδιότητε των, θεσμικών οργάνων και κάνουν πράγματα τα οποία έχουν ήδη απαγορευτεί. Και ίσως θα ήταν καλό να κοιτάξουμε την ανάγκη για αναθεώρηση της νομοθεσίας, φέρει στα θέματα των νάνο Είναι απαραίτητο να προβούμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι απαράδεκτο ε, να, είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν καθόλου έλεγχοι στη χρήση αυτών των νάνο σε τρόφιμα. Ε, ή των ποσοτήτων τους. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που είναι σαφείς πιστεύω για όλους εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρέπει ο καταναλωτή να είναι ενήμερος για την προέλευση των τροφίμων που καταναλώνει, εάν αυτά προέρχονται από κλωνοποιημένο ζώο ή από κατιόντες του. Χρειάζεται ανιχνευσιμότητα, χρειάζεται σήμανση. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η απο κατιοντε του χρειαζεται Δαλή έχει οτι η επιτροπο δαλη βούληση να ρίξει άπλετο φω στην υπόθεση αυτή και να δώσει απαντήσει στα πολυάριθμα εκκρεμή ακόμη σήμερα ερωτηματικά. Είναι αδύρυτη ανάγκη η ιχνηλασιμότητα ή ανεχνευσιμότητα για να μπορεί να επιλέγει έχοντας γνώση της καταστάσεως ο ε, καταναλωτής. Δεν μας, δεν ε, μας επιτρέπεται να ε, εκφράσουμε μια στάση η οποία θα ερμηνευτεί από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ως η Ευρώπη μένει αδρανή, η Ευρώπη δεν λαμβάνει αποφάσεις, η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνήσει. Θα πρέπει, κύριε Επίτροπε, να ξεπεράσετε την ε, θεσμική αυτή, το θεσμικό αυτό αδιέξοδο που διαπιστώθηκε για να δώσετε πιο πολλές εγγύσεις και στον καταναλωτή αλλά και στην ε, βιομηχανία των τροφίμων. Και τη γεωργική βιομηχανία θα πρέπει ως εκ τούτου να ε, κερδίσουμε το χαμένο έδαφος γιατί έχει περάσει πολύ καιρό και να τα προχωρήσουμε ταχύτητα σε ρύθμιση των ζητηματών. Ο κύριος Σαρσένης, ένα λεπτό. Αγαπητέ Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, εγώ θα είμαι λιγότερο διπλωματικός προτείνεται απαγόρευση από τα για τα κλωνοποιημένα τρόφιμα. Αλλά επίτροπε, κανένα δεν μπορεί να αγοράσει τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα. Τα κλωνοποιημένα ζώα είναι πολύ ε, ακριβά για να χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα. Αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα είναι οι κατιόντε του. Γι' αυτό θέλουμε απαγόρευση των κατιόντων. Θέλουμε σαφή σήμανση για του κατιόντε. Αλλά φοβούμε πω ο ρόλο σα στι διαπραγματεύσει δεν ήταν παραγωγικό εσείς ε, ήσασταν κατά της σήμανση των ε, κατιόντων. Ε, ήταν όμως ο ελάχιστος παρονομαστής συμφωνίας για το Συμβούλιο. Ήταν η μόνη μας επιλογή να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Παρακαλώ μάθετε τα διδάγματα, ακούστε τι έχουμε να πούμε εμείς για αυτό το θέμα και επανέλθετε με νέα αξιοπρεπή πρόταση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι και όλοι που με βαθύτατα που έχουν αποτύχει οι διαπραγματεύσεις και ιδιαίτερα καθώς έχουμε τώρα ε, να περιμένουμε μερικά χρόνια ακόμη μέχρι ότου προχωρήσουν ε, οι ρυθμίσεις για την τεχνολογία και την εισαγωγή των ε, προϊόντων από ζώα από τρίτα κράτη. Μέχρι να ρυθμιστούν όλα αυτά λοιπόν να πούμε ότι ε, αποτέλεσαν ένα σημαντικό σημείο αποτυχίας των προσπαθειών μας αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις. Νομίζω ότι ήταν ανάξιες της σημασίας ε, των, ε, του αντικειμένου τους. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και γι' αυτό τελικά απέτυχαν και οι διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να πω ότι συζητούμε για πολλά πράγματα, για πολλά ε, νομοθετήματα. Στη γενετική ε, μηχανική έχουμε επίση ακολουθήσει το ίδιο σύστημα. Δεν θέλουμε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Θέλουμε να έχουμε κάποιε οριακέ τιμέ. Θέλουμε να ε, έχουμε ασφαλή δεδομένα, εγγυήσει δηλαδή ασφαλεία. Εν τω μεταξύ έχει προχωρήσει η γενετική τεχνολογία και θα ήθελα να επισημάνω ότι τα κλωνοποιημένα ζώα δεν πληρούν καν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας σχετικής με την προστασία των ζώων, της ευημερίας των ζώων. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτή η πτυχή λησμονείται σιγά σιγά. Η γενική απαγόρευση δηλαδή της διάθεσης κλωνοποιημένων ζώων είναι για μένα αμφίβολης αποτελεσματικότητας και θα πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί τι είδους βάση μπορούμε να θεσπίσουμε ώστε να έχουμε σαφείς κανόνες και να μην προσπαθούμε μέσω της νομοθεσίας να παρεμποδίσουμε τις εξελίξεις και την επιστήμη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει η κυρία Σαρμπιού για 1,5 λεπτό. Εγώ να σας πω ότι αισθάνομαι απογοήτευση όσον αφορά την αποτυχία των ε, διαπραγματεύσεων διότι μήνες, χρόνια δουλεύουμε και τελικά δεν πετύχαμε τίποτα. Σε πάρα πολλά ε, σημεία τα είχαμε βρει και θα πρέπει να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Όσον τώρα αφορά τα ζωά που και τους κατιόντες τους θα πρέπει να είμαστε ελαστικοί. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουν οι Ευρωπαίοι. Δεν θέλουν κλωνοποιημένα ζώα και κρατιώντες τους κατά τις διαπραγματεύσεις. Το Συμβούλιο δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτά. Αυτό είναι καταδικαστέο. Εμείς κάνουμε υποχωρήσεις, δεχτήκαμε κάποια πράγματα τα οποία ήθελε το Συμβούλιο ακριβώ για να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να θεσπίζουμε δημοθεσία που να επιτρέπει τέτοια προϊόντα στο τραπέζι μα. Θα πρέπει τουλάχιστον να επισημαίνεται το περιεχόμενο εις την συσκευασία. Στην ετικέτα. Επίση, είχαμε πει ότι θα πρέπει να απογραφούν κάποιε τεχνικέ χρονοποίησει όσον αφορά την παραγωγή κάποιων ε, ειδών διατροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, να υπάρχει αυτή ανιχνευσιμότητα, ιχνηλασιμότητα για το, το, το, το, από πού προέρχεται ε, κάποιο τέτοιο είδος διατροφής ε, το οποίο προέρχεται από τρίτη χώρα. Επομένως θα πρέπει όλα αυτά να φύγονται από τη νέα πρόταση που θα προκύψει και θα πρέπει επομένω και τα κράτη-μέλη να προσέξουν περισσότερο αυτά τα οποία με θεμητό τρόπο προσδοκούν οι Ευρωπαίοι. Ευχαριστούμε εμεί, λέει πρώτα και τώρα η κυρία Γκαρντίνη για μισό λεπτό. Ε, Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι και εγώ ήμουν τμήμα τη αντιπροσωπεία για τη συνδιαλλαγή και πρέπει να πω πω τα ε, σήματά μα ήταν ε, ελπίδα, απογοήτευση αλλά και οργή. Ε, επιτρέψτε μου να πω γιατί εμεί εδώ ήμασταν ε, αντιπρόσωποι πάνω από 500, 500 εκατομμυρίων πολιτών. Είναι πολίτε που επαναλαμβάνουν με δυνατή φωνή ότι δεν θέλουν στη μεγάλη του πλειοψηφία να έχουν στα τραπέζι του τα τρόφιμα αποκλωνοποιημένα κλωνοποιημένα τρόφιμα, από κλωνοποιημένα ζώα, συγγνώμη, και από τους κατιόντε του Η σήμανση θα ήταν το μίνιμουμ. Είχαμε δεχτεί το μίνιμουμ. Αν είχαμε δεχτεί αυτή τη συμβαστική λύση, θα είχαμε δεχτεί μια κενή, ένα κενό ουσία ε, συμβιβασμό ε, Λίγο μακιγιάρισμα θα είχαμε κάνει, λίγο ε, καπνό στα μάτια των ανθρώπων. Για τα υπόλοιπα δεν υπήρχε καμία ρύθμιση. Θα είχαμε δεχτεί την απορρίθμιση και αυτό δεν ήταν δυνατόν. Δεν μπορούμε όμως σήμερα να είμαστε εδώ ακόμα μια φορά να υπερασπιζόμαστε τις επιλογές ε, αυτό που ήταν μια και να λέμε ότι ήταν συλλογική αποτυχία. Υπήρχε συμφωνία σχεδόν σε όλα και δυστυχώς αποτύχαμε και δώσαμε την εντύπωση στους πολίτες ότι οι μεγάλες βιομηχανίες και οι κανόνες του εμπορίου ε, αξίζουν πολύ περισσότερο από την, ε, πολιτική, ε, την ευρωπαϊκή ηθαγένεια την οποία εμείς υποστηρίζουμε εδώ. Γι' αυτό σας παρακαλώ ας ξεκινήσουμε μια νέα στάση, μια νέα αίσθηση γιατί θέλω και ελπίζω την επόμενη φορά οι προσδοκίες και η βούληση των πολιτών θα γίνουν σεβαστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκαρδίνη. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Μόρκου Νάιτε Μικουλένη. Κυρία Πρόεδρε, όλοι συμφωνούμε ότι η πληροφορία είναι αυτό το οποίο το πιο σημαντικό στον σύγχρονο κόσμο και αυτό ισχύει και για την ασφάλεια, την διατροφική. Οπότε όντως θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση όσον αφορά τα τρόφιμα. Αυτό ισχύει και για τους χυμούς των φρούτων. Όμως δεν καταφέραμε να βρούμε μια συμβαστική λύση όσον αφορά την ετικετοθεσία, ε, το, ε, ε, έτσι κάναμε πίσω γύρισμα επομένω. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος. Τώρα, βάλαμε τροχοπέδες επιχειρήσεις. Κάποια κράτη-μέλη ή σαν αντίθετα με αυτά τα οποία εμείς προτείναμε υπέρ των καταναλωτών, το ώστε να μπορεί ο κόσμος να δει από πού προέρχεται το γάλα το οποίο αγοράζουμε. Θα πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσον ε, θα χρησιμοποιούνται ε, οι νέες τεχνικές και νέες τεχνολογίες. Ελπίζω ότι θα γεφυρωθούν οι διαφορές μας. Περνάμε στη διαδικασία Κατσιδιάκη και δίνω το λόγο στην κυρία Μαγκίνης για ένα λεπτό. Ποιον έχει καταπλήξει ότι δεν καταλήξαμε συμφωνία. Εγώ τουλάχιστον ε, απ' έξω που τα έβλεπα, έβλεπα, διαπίστωνα πολλέ διαφορέ στην τράπεζα των συζητήσεων. Το να ξεκινήσει μια συνεδρία στι 7 το βράδυ και να καταλήξει να στεφθεί σε αποτυχ... με αποτυχία τη 7 το πρωί δεν ήταν και τόσο σπουδαία ιδέα στη τελευταία ανάλυση. Θα ήταν ε, λύση να χωρίσουμε τα νομοθετήματα σε δύο κομμάτια. Η κλωνοποίηση είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που πολλοί άλλωστε έθιξαν και νωρίτερα υπό τη σκοπιά τη ευημερίας των ζώων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να δούμε επίση και πώ με βάση του κανόνε του ΠΟΕ μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα της ε, χρήση της τεχνολογίας, γιατί θέλουν και οι γεωργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία στη θέση τους για να έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα. Άρα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα αυτά κατά τρόπον ε, ικανοποιητικά. Όσο δε αφορά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τη σύγκριση τους με αυτές που ισχύουν στον υπόλοιπο κόσμο, όταν εισάγουμε ε, προϊόντα κρέατος από τρίτα κράτη, είμαστε βέβαιοι ότι ισχύουν τις προδιαγραφές που έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαγκίνες. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κάτνα. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τον Επίτροπο για τις ε, προσπάθειές του στον τομέα της πρόληψης, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές πιστεύω και ιδιαίτερα όσον αφορά τα κλωνοποιημένα ε, υλικά ή υλικό από κλωνοποιημένα ζώα. Εγώ θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι να εκπροσωπώ τον Ευρωπαίο, την Ευρωπαία, που έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για πολύ προσεκτική στάση απέναντι στα κλωνοποιημένα προϊόντα. Θέλουμε κατά συντριπτικό ποσοστό όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, τουλάχιστον τη σήμανση για να μπορούμε να εντοπίζουμε ποια είναι τα προϊόντα από κλωνοποιημένο ζώο ανεξαρτήτως γενναίας. Και έχουμε επίσης, κύριε Επίτροπε, την απόλυτη δυναμία να καταλάβουμε γιατί το Συμβούλιο αντί ε, μέσω των ε, προφανώς εκλεγμένων επίσης μελών του, κυβερνήσεων δηλαδή, προτίμησε να υπηρετήσει τη συμφέροντα των αγορών και όχι των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Σουσλίνγκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε. Η πολιτική για την προστασία του καταναλωτή αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όταν λοιπόν καταφέρνουμε να εισάγουμε και να επιβάλλουμε αποτελεσματική πολιτική για τον καταναλωτή, ε, θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιου είδους αποτυχίες. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτύχαμε παταγωδός. Αν και θα ήθελα να επισημάνω ότι ορισμένοι προσπάθησαν ε, να προβάλλουν υποτίθεται, γιατί ξέρανε ότι θα προχωρήσουν σε αποτυχία, ε, τα λεγόμενα συμφέροντα των γεωργών και να επισύσουν τον κίνδυνο ενός μαζικού εμπορικού πολέμου με τους εμπορικούς μας εταίρους. Ελπίζω λοιπόν ότι έχετε το δυνατό επίτροπο θα καταθέσει νέα πρόταση για τα κλωνοποιημένα ζώα στην ε, Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο, πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αναλάβετε δράση και η απαγόρευση των κλωροποιημένων νομίζω αποτελεί μόνο ένα βήμα, ε, μόνο προσωρινό, γιατί εν τέλει χρειάζεται να έχουμε μια ουσιαστική νομοθεσία για το, που να ρυθμίσει τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζομπούρσκα. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να αναζητήσουμε την ίδια του προβλήματος. Το φταίχτη όμως μιλάμε για ένα θέμα στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία. Η Ντόλη το τελευταίο ζώο το οποίο κλωνοποιήθηκε. Χιλιάδε ζώων πέραν από αυτή τη διαδικασία. Φινησιγενή, παραμορφωμένα ζώα έχουμε. Πρόκειται για βασανισμό εις βάρος αυτών των ζώων. Επομένω, θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση μέσα αυτής της οδηγίας ε, για τους κατιόντες των ζώων αυτούς, για το, το κρέας τους. Θα πρέπει να στείλουμε σήμα. Το μήνυμα να είναι ότι τέτοιου ζώα θα πρέπει να κυκλοφορούν για να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, τα αποκαλούμενα νέα τρόφιμα είναι προϊόντα και ε, ε, τροφικά συστατικά που έχουν υποστεί αλλαγή της ε, τροφικής τους αξίας. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες για την νομοθεσία αυτή. Ποια θα είναι η σχέση με την νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς εφόσον η κλωνοποίηση είναι τμήμα της γενετικής μηχανικής και προέρχονται από γενετική τροποποίηση ρυθμιστεί, πώς θα ρυθμιστούν αυτά τα τρόφιμα στα διάφορα κρατημέλη, πώς θα γίνονται τα, οι έλεγχοι για την ασφάλεια αυτών των νέων τροφίμων, ποια θα είναι τα κριτήρια για τον ορισμό αυτών των προϊόντων και κυρίως και πάνω απ' όλα πώς θα ενημερώνει το καταναλωτής για τα χαρακτηριστικά και τις ε, τροφικές ιδιότητες των νέων τροφίμων που θα αγοράζει. Αυτό το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές είναι η προστασία του καταναλωτή και η ασφάλεια των τροφίμων στη χρήση των νέων αυτών προϊόντων και άρα σωστή ενημέρωση του καταναλωτή. Γι' αυτό και πιστεύω πω η ανιχνησιμότητα, ιδιαίτερα των φυσικών προϊόντων που ήδη έχουμε δυσκολία να το κάνουμε, να είναι απόλυτη και πλήρη για τον καταναλωτή. Ευχαριστούμε κύριε Σκοτά και τέλο το λόγο έχει η κυρία Τζαβέλα. Το όλο θέμα πιστεύω ότι προήλθε από τη μη ενημέρωση των καταναλωτών και των πολιτών. Όταν υπάρχει αδιαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών της Ευρώπης και όλου του κόσμου. δημιουργούνται αδιέξοδα και δεν καταλήγουμε κάπου. αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι όταν βλέπετε ότι υπάρχει ισχυρή αντίδραση για προϊόντα από καντιόντα, θα έπρεπε και εμείς και οι αποφασίζοντες και νομοθετούντες να υπακούουν στο πνεύμα το οποίο απαιτεί η κοινή γνώμη. ενημέρωση λοιπόν και διαφάνεια σε ό,τι κάνουμε για να μπορούμε να τελειώνουμε αυτό το οποίο αρχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Τζαβέλα. Έτσι τελειώνει η διαδικασία Catch the Eye και δίνω το λόγο στον κύριο Νταλή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ πάρα πολύ προσεκτικά σημείωσα όλα αυτά τα οποία εκφράστηκαν κατά την ε, συζήτηση. Οπότε ευχαριστώ του εξωτερικού βουλευτέ για τι απόψει του και θα σα διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί σα και όλου του εμπλεκόμενου. Και ο κοινό μα στόχο υπάρχει είναι το να προχωρήσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα και με τι δύο αυτέ προτάσει και για την κλωνοποίηση, τα κλωμμένα τρόφιμα και για τα νέα τρόφιμα και θα πρέπει επίσης να σας τονίσω το τι θέση ετηρήσαμε κατά την διαδικασία της συνδιαλλαγής. Και όπως προείπα, αυτό το οποίο έγινε ήταν το να αναζητούμε λύσεις, συμβιβασμούς, πράγματα ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Δικαιολογημένα και να διέπονται από αναλογικότητα. Ό,τι θα θέλαμε όλοι μας να δούμε. Και εγώ, σαν αρμόδιος για την πολιτική για τους καταναλωτές, ε, φυσικά και θέλω να υπάρχει ενημέρωση του καταναλωτή, όμως θα πρέπει όλα αυτά να είναι τεκμηρωμένα και θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας μια μελέτη αξιολόγησης για να διαμορφώσουμε τη θέση μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδέποτε είπε ε, ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τικετοθεσία. Όμως, πάσα απόφαση θα πρέπει να αξιολογείται για να μπορούμε να ξέρουμε τι αντικτύπο θα έχει επί των Ευρωπαίων καταναλωτών είτε παραγωγών είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε αυτή τη θέση και σας διαβεβαιώ ότι οι υπηρεσίες μας και ο υποφαινόμενος θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση όσο γίνεται. Όχι, δεν αναβάλλω τη λήψη αναγκαίων αποφάσεων. Η πρόεδρο. Κύριε Νταλή, σα ευχαριστούμε. Εξ ονόματο του Συμβουλίου, η κυρία Γκέρι, μέσω του εκπροσώπου τη, ο οποίο την αντικαθιστά γιατί έχει χάσει τη φωνή της σήμερα. Έχεις. Επίτροπε. ό,τι με κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα καταρχά να εκπροσωπήσω τι ευχαριστίε μου για τη συζήτηση εκ μέρους της Προεδρίας αλλά και εκ μέρους του Συμβουλίου και ιδιαίτερα θέλω να εκφράσω ε, τις ευχαριστίες μου σε όσους ε, τοποθετούμε μέσα στο Συμβούλιο εξέφρασαν ε, την ανάγκη να προχωρήσουμε σε νέα προσπάθεια για νομοθεσία. Στη διαδικασία για τη συνδιαλλαγή προβλήθηκαν πολλά επιχειρήματα που ακούστηκαν και εδώ. Θα θέλαμε επίσης να απορρίψουμε ε, υπενιγμούς ε, ότι είτε το Συμβούλιο είτε η Ουγγρική ε, Προεδρία υπήρξαν ανέντιμοι ή εξυπηρέτησαν συμφέροντα ιασδήποτε ομάδας πιέσεως. Μία από τις κύριες πτυχές ε, της συνθήκης Λισαβόνας είναι ότι ενισχύει την τον καταβερισμό ευθυνών. Ε, εμείς συνεχίσουμε την προσπάθεια από τη δική μας πλευρά, από το δικό μας μετερίζει, με την ελπίδα ότι θα φτάσουμε τελικά σε μια συμφωνία. Θέλουμε να μην υπάρχει βεβαιότητα ως προς το τι φαγητά φτάνουν στο τραπέζι μας. Κλωνοποιημένα ζώα ή προϊόντα αυτών προς το παρόν θα απαγορευθούν. Και θέλουμε να υπάρχει θα απαγορευθούν. Και θέλουμε να υπάρχει αριθμευσιμότητα για τους κατιόντες και σωστή σήμανση. Λύσεις υπάρχουν. Λογικέ λύσει. Όπω αυτό που έχει γίνει με το σαλάμι και αντίστοιχα προϊόντα. Θέλουμε λοιπόν τι λύσει που έχουμε στη διάθεσή μα να τι αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και θα ήθελα να πω προς την κυρία Λιωτάρη, η οποία επικαλέστηκε ένα ιστορικό έγγραφο του Συμβουλίου, ότι συζητήσαμε βέβαια τα θέματα αυτά και μας οδήγησαν στην κυρία μας θέση. Εσείς, παραθέτοντας από το κείμενο αυτό, επιλέξετε μία μόνο πρόταση και διαβάσατε. Παραλείψετε όμως το κομμάτι εκείνο της νομάτευσης που λέει ότι υπάρχουν κίνδυνοι σε σχέση με τους καρονές της ΠΟΕΜ. ή τα συμπεράσματα του γνωμάτευσης που λένε ότι η σήμανση μόνο θα αποτελούσε μια αποδεκτή λύση. Άρα ήταν μερική η παρουσίαση της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά όμως συμφωνώ μαζί σας ότι πριν να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Και με βάση αυτά θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Ως στην ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε πρόοδο. Ο κύριος Δαλή υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει χωριστή πρόταση για τα προϊόντα από ζώα, πράγμα το οποίο θεωρούμε καλό ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. Για την ολοκλήρωση της συζήτησης, τώρα ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Διαπραγμάτευσης στη Συνδιαλλαγή. Ο κύριο Πιτέλα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι από όλε τι παρεμβάσει των συναδέλφων, του οποίου όλου ε, ευχαριστώ, ξεκινώντα από την εισηγήτρια και από την ε, τεκμηρίωση που μας εξέθεσε η ίδια η στην οποία υπογραμμίζεται πως η απαδοχή των προτάσεών μας δεν θα οδηγούσε σε οποιοδήποτε εμπορικό πόλεμο. Όλα αυτά απέδειξαν και το λέω χωρίς διάθεση εναντίον, το λέω προς την Ουγγρική Προεδρία. Όλα αυτά που δείχνουν ότι δεν υπήρξε συλλογική αποτυχία. Η αποτυχία υπήρξε αλλά αφορά ένα ε, μέρος και πρόκειται για σαφή ευθύνη των κυβερνήσεων. Τώρα, πέρα από αυτό και μην μου πείτε ότι η απλή σήμανση του βοηού κρέατος των κλωνοποιημένων ζώων ούτε καν των κατιόντων θα μπορούσε να θεωρηθεί μια αξιοπρεπής και ικανοποιητική συμφωνία για το Κοινοβούλιο γιατί ήταν λίγο πάνω από το μηδέν αυτή η συμφωνία και τώρα τι κάνουμε. Τα ξεχνάμε όλα αυτά και προχωράμε μπροστά. Και κυρίως ζητάμε από το Συμβούλιο να ζητήσει να συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις. Ξέρετε ποιες είναι οι θέσεις του Κοινοβουλίου και οι θέσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Σήμανση των προϊόντων των κλωνοποιημένων ζώων και των κατιόντων τους. Αυτό είναι το μίνιμουμ. Δουλέψτε εκεί με τις κυβερνήσεις να δεχτείτε αυτό το μίνιμουμ. Και έπειτα, Επίτροπε Ντάλη, εγώ ξέρω πως εσείς ε, έχετε πολύ καλή βούληση και ας μας παρουσιάσετε όσο γίνεται πιο σύντομα τον τρόπο ώστε να επιτρέψετε σε αυτό το κοινοβούλιο να εγκρίνει την νομοθεσία για την κλωνοποίηση. Η μία πρόταση που να κάνει δεκτές τις προτάσεις μας και έπειτα προχωρήσουμε και για τα νανοηλικά. Αν βγάλουμε το τμήμα της κλωνοποίησης από εκεί μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Τελευταία παρατήρηση και όλοι διαπιστώσατε την ενότητα του Ευρωκοινοβουλίου. Πολύ σημαντική ενότητα. 360 μοίρες συμφωνίε. Ίσως και να κάνατε κάποιο λάθος στι διαπραγματεύσει όταν σκεφτήκατε ότι δεν υπήρχε τέτοια συμπαγή θέση από πλευρά του Κοινοβουλίου. Μην το κάνετε πια αυτό το λάθος για τα λεπτά ζητήματα που αφορούν την υγεία των πολιτών. Είμαστε και θα είμαστε ενωμένοι. Point d'ordre, Monsieur Τέλος της συζήτησης. Κύριε Στάς, τι θέλετε διαδικαστικό. Ε, στη διάρκεια αυτής της συζήτησης ε, επανειλημμένως αναφέρθηκε η στάση του κυρίου Ντεκούχτη και επίσης ε, ετέθη μια ερώτηση προς τον κύριο Νταλή για το κατά πόσο γνώριζε την νομική θέση γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Κύριε Νταλή, άκουσα την απάντησή στις ερωτήσεις σας, αλλά σε αυτή την ερώτηση δεν απαντήσατε και είναι πολύ σημαντική η ερώτησή μας. Η έλλειψη συμφωνίας μέσα στην Επιτροπή αν υπάρχει, θα ήταν ε, ε, κέρια σημασία. Ο ε, κύριος Δεγκούχτο φαίνεται να... Έχει χρησιμοποιήσει λάθος επιχειρήματα. Θέλω να ξέρω ποια είναι η απάντησή σας λοιπόν. Εν μέρει αποφυθήκατε στην εισηγήτρια για αυτήν την ερώτηση. Θα ήθελα να προτείνω στον Επίτροπο να απαντήσει. Θα πρέπει να προσέχετε Όμω, γιατί εγώ πιστεύω πως απάντησε, θα κλείσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση και θα περάσουμε στην επόμενη. The uh, next item on the agenda is the Επόμενο θα μας ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προ τον και την Επιτροπή για την επανεκτάση πρωτοβουλία σχετικά με τις ΜΜΕ, Small Business Act.